Hanno votato άπαντες. Υπάρχουν ακόμα βουλευτές που πρέπει να ψηφίσουν. Οι ψηφολέκτες ψήφισαν ε, και οι ίδιοι. Υπάρχουν ακόμα βουλευτές που πρέπει να ψηφίσουν. Από τις κάλπες μου ζητάνε 5 λεπτά χρόνο. εντάξει. okay. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα τη ψηφοφορία και καλό του ψηφολέκτε να πάνε στην αίθουσα R15 για να μετρήσουν τις ψήφους. Η έναρξη της συνόδου ξανά θα ανακοινωθεί στις οθόνες και με τα κουδουνάκια.